Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, το σημερινό αποτέλεσμα έδειξε ότι η πλειοψηφία ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, αντί να προχωρήσει στην δημοκρατία θέλει να μείνει μεταξύ τους. Το 2014 μια απόφαση στη, δημοκρατία, στη Γερμανία έδειξε ότι θέλουν να συμμετέχουν, αλλά στο μέλλον δεν μπορούν να κινούνται, δεν μπορούν να εκφράζονται. Και ε, όλο και περισσότερο αυξάνεται η απαξίωση. Ο συνάδελφος Γιώλα Λάινεν των σοσιαλιστών ε, μας προειδοποίησε για αποσταθεροποίηση λόγω μικρών κομμάτων. Στη Γερμανία ήρθαν 7 ε, βουλευτές από μικρά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί καταργήθηκε το αντιδημοκρατικό κατόφλι. Μα είναι 751 όλοι οι βουλευτές, οι 7 θα σας αποσταθεροποιήσουν ε, ή θα ε, πλήξουν ή θα περιορίσουν τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου. Το δικό μου κόμμα, το Εθνικιστικό Κόμμα της Γερμανίας N5, θα αντισταθεί και θα μετέλθει κάθε νόμιμου μέσου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Δεν ήθελα να μιλήσουμε για τα εκλογικά συστήματα στην Ευρώπη και τις μεταρρυθμίσεις. Ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Πόσπισίλ, αλλά ε, αποσιάζει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 σε κάθε κρατήδιο υπήρχε, επικρατούσε διαφορετικό εκλογικό σύστημα και όταν ο Χίτλερ πήρε την εξουσία εναρμόνισε όλα τα εκλογικά συστήματα. Είναι μια παλιά μεθοδός που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθεί το υπόδειγμα του Χίτλερ για να τα ισοπεδώσει όλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαλυθεί. Η Πρόεδρος, πολύ σύντομο ήταν αυτό. Μπορεί να έχετε τύχει να βρείτε και κανένα ταξί φεύγοντας. Ο Άντερσον. Υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία απαξίωση και μία δυσφορία. Ε, οι βουλευτές εκλέγονται από τους πολίτες της χώρας τους. Ε, ε, οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να εκλέγονται από ένα ευρωπαϊκό μανιφέστο. Αλλά καμιά φορά αυτό σημαίνει τεχνητή υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Αυτή η πρόταση με τα εθνικά, διεθνή μάλλον και ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια και λίστες που θα κατεβάζουν ε, τα ευρωπαϊκά κόμματα και να έχουν και το λογότυπό τους στο ψηφοδέλτιο. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Εκχωρούνται ε, εξουσίες από τα ε, ευρωπαϊκά κράτη στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και αυξάνεται έτσι η απόσταση μεταξύ των εκλογέων και των εκλεγμένων εκπροσώπους. Ελπίζω αυτές οι ε, κακές προτάσεις να μην ευδοκιμήσουν. Η ο κύριος Μπάλτσο. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι καταψήφισα τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω και για ποιο λόγο. Ε, εντολή του Ευρωπαίου Βουλευτή ε, απορρέει από διαφορετικά εκλογικά συστήματα. Υπάρχει κριτική στην Ευρώπη και απέναντι στην πολυμορφία της. Ευτυχώς δεν την έχουμε απεμπολίσει εντελώς. Ε, η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει τόσο ενιαία ε, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό και ελπίζω ποτέ να μην συμβεί. Η πρόταση φιλοδοξεί στο να υπάρχουν κοινέ εκλογικέ περιφέρειες, ενιαία ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια. Τι άλλο θα δούμε δηλαδή. Και τα ευρωπαϊκά κόμματα να έχουν και τους επικεφαλής τους αρχηγούς τους, που να διορίζονται κεντρικά. Έτσι, υποσυνείδητα διαλύονται τα κράτη-μέλη και καταργούνται. Η πρόεδρος, ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω και εγώ για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να θυμίσω ότι είχα ζητήσει το λόγο και για το προηγούμενο, για τη μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές και δεν μου δώσατε το λόγο και δεν μπόρεσα να κάνω την αιτιολόγηση ψήφου μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μεταρρύθμισή του, υποστήριξα την ε, εισηγήτρια Χιούμπνερ και τον εισηγητή Λάινεν. Έχουν αλλάξει καιροί από την τελευταία φορά και από την τελευταία πρόταση. Είναι πάρα πολύ διαφορετική η σημερινή πρόταση και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ισότητα των φύλων στα ψηφοδέλτια. Αυτό δεν με ικανοποιεί. Υπάρχουν όμως άλλα καλά σημεία, όπως η ηλικία των 16 ετών για το δικαίωμα του εκλέγην ή η ηλεκτρονική ψήφος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, μην κάθεστε. Γιατί έχετε άλλη μια δήλωση ψήφου, επεξήγηση ψήφου για το μελλοντικό ε, πακέτο για την ε, αεροπλοεία. Σας δίνω το λόγο και πάλι. Είστε ο πιο ανθεκτικός βουλευτής απόψε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και για τη μελλοντική δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να κάνω την επεξήγησή μου προφορικά Υποστήριξα αυτό το κείμενο, μεταξύ άλλων, διότι σε λίγα χρόνια οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν ε, περικόψει πάρα πολλές θέσεις εργασίας, πάνω από 2.000. Ε, θα πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται εκεί και πώς εξελίσσεται αυτός ο κλάδος της οικονομίας. Τα λέει αυτά η έκθεση πολύ ωραία. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ε, μειώσουμε και το περιττό βάρος. Όχι βέβαια να κάνουμε εκτόσεις στην ασφάλεια, μόνο αλλά στη γραφειοκρατία υπάρχει χώρος για περικοπές. Υποστήριξα την έκθεση και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω την επεξήγησή μου. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα συνοπτικά πρακτικά της παρού συνεδρίασης θα εγκριθούν ε, στην επόμενη συνεδρίαση και αν δεν διαφωνεί κανείς.